Για την ενεργειακή απόδοση. Έχουμε 67 επεξηγήσεις ψήφου, 67 εγγεγραμμένους στον κατάλογο, θα πάει πάνω από μια ώρα δηλαδή. Γι' αυτό θα είμαι πολύ αυστηρό στην τήρηση χρόνου. Κυρία Ζανίκη, ένα λεπτό. Σιγά.